Τα άλλα εμεί καταγγέλουμε για δεύτερη φορά εμεί φέτο εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σα ευχαριστώ. Πριν συνεχιστεί η συζήτηση, θα ήθελα να καλωσορίσω μια αντιπροσωπεία της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου του Μεξικού υπό την ηγεσία της ε, κυρίας Γκαμπριέλα Κουέβας που είναι στη Γερουσία. Η αντιπροσωπεία επισκέφτεται διάφορα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και είχε ανταλλαγή απόψεων με τα μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου. Θα ήθελα ονόματι σας να τους καλωσορίσω για αυτή την επίσκεψη των εκπροσώπων του Κοινοβουλίου του Μεξικού που είναι σημαντικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και ισχυρός οικονομικός ε, εταίρος και φορέας στο παγκόσμιο προσκήνιο. Καλώς ήρθατε λοιπόν. Ευχαριστώ. Συνεχίζουμε. Η κυρία Κέλλερ έχει το λόγο για 1,5 λεπτό. Και πάλι απασχολούμαστε ε, μετά από μια προηγούμενη συνάντηση με τις συνδίκες εργασίας στην, στο και με τους νεκρούς που προκλήθηκαν από βιομηχανικές δραστηριότητες. Η κατάσταση είναι καταστροφική στο Μπαγκλαντές μέσα στο συνολικό σύστημα της κατανομής εργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο και μέσα σε μία φόρα στι συνθήκες εργασίας δεν πρέπει να μας εκπλήσει το ότι συμβαίνουν τέτοιες τραγωδίες. Προφανώς πρέπει η κυβέρνηση του Μπαγκλαντές να βελτιώσει την κατάσταση των εργαζομένων εκεί. Πρέπει να αυξηθεί ο κατώτατος μισθός, αλλά αυτό από μόνο του δεν φτάνει. Θα πρέπει να καταβάλλεται, θα πρέπει να μπορούν να εργάζονται οι εργατικές ενώσεις χωρίς καταστολή. Θα, να υπά... θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα προσφυγής στη δικαιοσύνη. Αυτό όμω το οποίο μπορούμε να κάνουμε εμεί ω Ευρώπη θα πρέπει επιτέλους οι επιχειρήσεις να αναλάβουν την ευθύνη τους. Θα πρέπει να τηρούν τις συμφωνίες που έχουν υπογράψει. Είναι κάτι το οποίο είναι ενοχλητικό και εξοργιστικό ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις παραγνωρίζουν αυτές τις συμφωνίες. Θα πρέπει να έχουν και την υποχρέωση να αποζημιώνουν τα θύματα αυτών των τραγωδιών και να πληρώνουν και το κόστος της νοσηλείας τους. Θα πρέπει να τηρηθούν οι ε, διεθνείς συμφωνίες. Υπάρχουν ορισμένες επιχειρήσεις οι οποίες εξασφαλίσουν ότι υπάρχει και έλεγχος των δραστηριοτήτων τους στα πλαίσια του δίκαιου εμπορίου. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να υποχρεώσει όλους να ακολουθούν μια τέτοια διαδικασία και αυτό μπορεί να γίνεται με τήσεις εκθέσεις ή με ετικετοθεσία στις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν θετικές πρακτικές. Και τέλος θα πρέπει να εφαρμοστούν όλες αυτές οι ρήτρες ως υποχρεωτικές και όχι να θεωρηθούν ότι μπορούν απλώς να αποτελούν ένα τμήμα της ε, αηφόρου αναπτύξεως και είναι θελοντικά. Πρέπει να εξασφαλίσουμε λοιπόν ότι θα γίνεται ένας αυστηρότερος έλεγχος και μια πιο διάφανη παρακολούθηση των εμπορικών δραστηριοτήτων των ευρωπαϊκών εταιριών με αυτούς τους προμηθευτές. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Συνάδελφε Λαγιαρίκη, έχετε το λόγο για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος δεν συγκλονίστηκε στο θέμα των 1200 θυμάτων της Ντάκα. Όλα αυτά θυμίζαν ένα στρατητικό νεκροταφείο. Οι άνθρωποι αυτοί έχασαν τη ζωή τους όχι λόγω ενός ατυχήματος, αλλά λόγω ενός εμπορικού πολέμου υπέρ των συμφερόντων των μεγάλων εταιριών για να εξυπηρετήσουμε τα συμφέροντα της βιομηχανίας του ενδύματος, θυσιάζοντας σκλάβους στο Μπαγκλαντές οι οποίοι δουλεύουν για 30 ευρώ το μήνα 12-15 ώρες την ημέρα. Τα κροκοδιλιά δάκρυα δεν αρκούν. Πρέπει να κάνουμε κάτι, να γυρίσουμε την πλάτη στην λατρεία της υπεραξίας των μεγάλων πολυεθνικών εις βάρος ανθρώπων. Πρέπει να επαναδιατυπώσουμε την εμπορική μας πολιτική, γυρώντα την πλάτη σε αυτήν την δραματική κατάσταση θεμελιώνοντας την συνεργασία μας σε νέες βάσεις. Λαμβάνοντας υπόψη ακριβώς τις βελτιώσεις που μπορούμε να επιφέρουμε στον τομέα της ασφάλειας, στη βελτίωση των μισθών και δίνοντας τη δυνατότητα στους εργαζόμενους στον Μπαγκλαντές να σχηματίζουν τα δικά τους συνδικάτα και να, μείνονται, να υπερμείνονται των συμφερόντων τους. Σας ευχαριστώ. Η ε, κυρία Κιώστιγκερ έχει το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Τα τρομερά νέα της τραγωδίας των Μπαγκλαντές μας έχουν συγκλονίσει όλους. Έχουν χάσει τη ζωή τους πάνω από 1.100 άνθρωποι και αυτό είναι μια τραγωδία για τις οικογένειές τους αλλά και για όλο τον Μπαγκλαντές. Αλλά θα πρέπει να ξέρουμε ότι αυτό έγινε γιατί δεν τηρήθηκαν οι προδιαγραφές ασφαλείας των κτίριων. Δεν είναι θέμα λοιπόν νομικών προδιαγραφών, αλλά είναι η έλλειψη ελέγχου. έχουμε ως αντίδραση καταφέρει να πείσουμε 40, πάνω από 40 εταιρείε να υπογράψουν μια συμφωνία με μη κυβερνητικέ οργανώσει και άλλου φορεί για τη βελτίωση τη διαδικασία παραγωγή. Αυτό είναι ένα θετικό και σημαντικό βήμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις επιχειρήσεις της, γιατί δεν αρκεί να δημιουργούν θέσεις εργασίας στις αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά θα πρέπει να δίνουν και το μήνυμα των ευρωπαϊκών αξιών. Η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η βελτίωση των συνδικών εργασίας, η τήρηση των προδιαγραφών του περιβάλλοντος και η δημιουργία ευμάρειας στις χώρες παραγωγής πρέπει να είναι ο στόχος μας. Μέσω του γενικευμένου συστήματος προτιμήσεων η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τη δυνατότητα να εξασφαλίσει ότι και η εμπορική της εταίροι και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αναλαμβάνουν την ευθύνη για τις διαδικασίες αυτές της παραγωγής. Το Μπαγκλαντές είναι δεσμευμένο να τηρεί τις ε, συμβάσεις του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας και του ΟΗΕ. Πρέπει όμως να εξασφαλίσουμε ότι και ο τελικός καταναλωτής θα δεσμεύεται ότι θα πρέπει να κατανοεί ποιες είναι οι συνθήκες εργασίας στις χώρες παραγωγής και να αποδέχεται ή όχι τα προϊόντα αυτά. Πρέπει να υπάρξει λοιπόν μεγαλύτερη διαφάνεια για τα θέματα αυτά. Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να γνωρίζουμε τα προϊόντα αυτά τα οποία έρχονται στην ευρωπαϊκή αγορά αν τηρούν τις προδιαγραφές του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας ή όχι. Η συμφωνία αυτή με τις, ε, των εταιριών με τους παραγωγούς ενδυμάτων δίνει τη δυνατότητα ο καταναλωτής να έχει περισσότερη πληροφορία και έτσι να εξασφαλίσουμε ότι θα γίνει η παραγωγή σε αηφόρο τρόπο με τις κατάλληλες αποδοχές και με τις προδιαγραφές ασφαλείας. Αυτό πρέπει να είναι ο στόχος αυτής της εφαρμογής της συμφωνίας που ανάφερα προηγουμένως. Ευχαριστώ. Κύριε Κέστιγκερ, δεχόσαστε μια γαλάζια κάρτα. Γαλάζια κάρτα. Υπάρχει γαλάζια κάρτα για σας. Ναι, ορίστε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Κιώστιγκερ, θα ήθελα να σας ρωτήσω όπως και άλλους για κάτι το οποίο δεν νομίζω ότι έχει τονιστεί ιδιαίτερα στη συζήτηση αυτή. Ήταν μια τρομερή τραγωδία που έγινε στο Μπαγκλατές με πάνω από χίλιους νεκρούς. Όλοι νιώθουμε ότι είναι σκανδαλώδες αυτό. Αλλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτά γίνονται και περνάνε και μετά από μια εβδομάδα όλοι έχουμε ξεχάσει. Μήπως θα πρέπει να προχωρήσουμε σε μέτρα τα οποία να είναι μη αντιστρεπτά και να αποτρέψουν την επανάληψη αυτών των γεγονότων όχι μονάχα στο Μπαγκλαντές αλλά στη Κίνα, στη Σιγκαπούρη, την Κορέα και σε άλλες ασιατικές χώρες όπου δεν υπάρχουν ούτε οι ελάχιστες συνθήκες ασφάλειας των εργαζομένων, ούτε οι κοινωνικοί, κοινωνικές προδιαγραφές για την εργασία. Μήπως λοιπόν το καλύτερο μέσο για να το πετύχουμε αυτό είναι να εξασφαλίσουμε ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα μπορούν να υφίστανται κυρώσεις σε τέτοιες περιπτώσεις ώστε να τις ε, εμποδίσουμε να παράγουν προϊόντα σε τέτοιες συνθήκες. Υποστηρίζετε ένα τέτοιο μέτρο. Νομίζω ότι αυτό το οποίο θέτεται ως ερώτημα είναι φυσική συνέπεια της συζήτησής μας σήμερα. Προφανώς θα πρέπει να βελτιώσουμε όλες αυτές τις ε, συνθήκες ώστε τα ατυχήματα που έγιναν στο Μπαγκλαντές και στην Καπότσι να μην επαναληφθούν. Γιατί αυτά δεν έγιναν γιατί υπήρχαν ε, ελλειπείς νομοθετικές ρυθμίσεις αλλά επειδή δεν τηρήθηκαν όλες αυτές οι προδιαγραφές. Πιστεύω ότι εδώ θα πρέπει να ασκήσουμε πίεση ώστε να υπάρξει σωστή εφαρμογή και δεν είναι μονάχα οι αλυσίδες φτηνής παραγωγής οι οποίες χρησιμοποιούν τέτοιες ε, εγκαταστάσεις αλλά και μεγαλύτερες εταιρείες και εδώ θα, μπορούμε να πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες να ασκήσουμε πίεση σε αυτές τις μεγάλες εταιρείες. Σας ευχαριστώ. Κύριος Μωρέρα έχει το λόγο για 1,5 λεπτό. Ε, ε, Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, εδώ και λίγους μήνες ήταν η τραγωδία στο εργοστάσιο ενδυμάτων στο Μπαγκλαντές και τώρα έχουμε ένα νέο τρομερό ατύχημα, μια τραγωδία που έγινε στην ίδια χώρα με το θάνατο πάνω από χίλιων εργαζομένων στην ΤΑΚ λόγω της κατάρρευσης ενός κτηρίου όπου γινόταν παραγωγή ενδυμάτων. Εγώ χαιρετίζω βέβαια τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν από το Μπαγκλαντές και επίσης και τα μέτρα που έλαβαν ορισμένες ευρωπαϊκές εταιρείες για να εξασφαλίσουν ότι θα τηρούνται οι ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας στα πάνω από 5.000 εργοστάσια του Μπαγκλαντές. Το θέμα όμως είναι να εφαρμοστούν αυτά στην πράξη. Οι εταιρείε θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι πράγματι θα τηρηθούν αυτές οι, οι ευθύνε που έχουν σε κοινωνικό και επιχειρηματικό επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως δεν μπορεί να δίνει στο Μπαγκλαντές την ευνοϊκή εμπορική μεταχείριση σε επίπεδο εμπορίου αν οι χώρες αυτές συνεχίσουν να παραβιάσουν συστηματικά τις πιο στοιχειώδες υποχρεώσεις που έχουν. Δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να δέχεται ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις χωρίς συνδυασμούς εκμεταλλεύονται τις άθλιες συνθήκες εργασίας στο Μπαγκλαντές και παρόλα αυτά να συνεχίζουν να λειτουργούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να εισάγουν προϊόντα τα οποία έχουν παραχθεί με κόστος ζωές σε χώρες όπως το Μπαγκλαντές. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Συνάδελφε Ντέλη, έχετε το λόγο για ένα λεπτό. Αγαπητοί συνάδελφοι, πάνω από 1.100 νεκροί. Αυτός είναι ο μακάβριος απολογισμός που χρειάστηκε για να δείξει τον ενδιαφέρον της επιτέλους στη διεθνή κοινή γνώμη. Χρειάστηκε μια καταστροφή στο Ραζαπλάζα για να κινητοποιηθούμε. Αλλά θα σας δώσω και άλλα νούμερα. 20 ευρώ για ένα παντελόνι, μια φούστα, κάποια συγκεκριμένη μάρκα. Κυρίε και κύριοι, έω πότε οι εργάτε τη Ασία θα γίνονται θύματα εκμετάλλευση στα πλαίσια τη χειρονή δουλεία κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί. Υποτίθεται ότι κάποιε εταιρείε υπέγραψαν συμφωνία για να βελτιωθούν οι συνθήκε εργασία. Αλλά αυτό δεν αρκεί. Πρέπει να τροποποιήσουμε την ευρωπαϊκή νομοθεσία, ώστε οι μητρικέ εταιρείε να είναι υπεύθυνε για τι πρακτικέ των υπεργολάβων του. Πρέπει να σταματήσουμε επίση τη μεταφορά τη παραγωγή προ χώρε όπου οι συνθήκε εργασία είναι πολύ χειρότερε το είπαν και οι συνάδελφοι, πρέπει επίση ο συνδικαλισμός να είναι ελεύθερος και αυτοί οι άνθρωποι να ζήσουν αξιοπρεπώς χάρη στου μισθού του. Μην ξεχνούμε όμω ότι η εταιρική κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων πρέπει να συμπεριλάβει και το περιβάλλον. Οι επιχειρήσεις αυτέ δυστυχώ αγνοούν και το περιβάλλον και το ξεχάσαμε και εμεί σε αυτήν τη συζήτηση. Ένα τέλος λοιπόν στην απώλεια ανθρώπινων ζώων σε όλο τον κόσμο. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Μάιερ έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Λέγεται στο κεφάλαιο ότι το κεφάλαιο ενδιαφέρεται μόνο για το κέρδος. Αν μπορέσει να έχει κέρδος, μπορεί να ανανεώνεται. Στο 20% αρχίζει να γίνεται παραρμητικό. Στο 50% αρχίζει να παραβιάζει όλους τους κανόνες και όταν φτάσει στο 300% το κέρδος δεν οροδεί προ ουδενός εγκλήματος. Αυτό είναι ακριβώς το πρόβλημα. Το ευρωπαϊκό κεφάλαιο είναι συνυπεύθυνο για αυτό το έγκλημα. Είναι συνυπεύθυνο ένα σύστημα το οποίο είναι απάνθρωπο και διεφθαρμένο και βασίζεται στην απορρίθμιση στους φορολογικούς παραδείσους και στην μετακίνηση των επιχειρήσεων σε φτωχότερες χώρες. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της νεοφιλελεύθερης Ευρώπης γιατί το μόνο πράγμα το οποίο ενδιαφέρει τις επιχειρήσεις είναι η συσσόρευση κεφαλαίου σε βάρος των ε, ανθρωπίνων ζωών, σε βάρος της ευρωπαϊκής ένδυας. Δεν υπάρχει κανένας ενδιασμός για να μπορέσουμε να συσσωρεύσουμε κεφάλαιο, κεφάλαιο, περισσότερο κεφάλαιο. Ευχαριστώ κυρία Σαΐφη για δύο λεπτά. Merci. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, όπως και οι συναδελφοί, να εκφράσω καταρχήν τα συλληπιτήριά μου στα θύματα του Ραναπλάζα. Αλλά δεν είναι μόνο τώρα πλάζει. Είχαμε και τα πρόσφατα ατυχήματα στην Καμπότζη. Όπως είπα και τον Ιανουάριο, το παραλαμβάνω σήμερα, οι επιχειρήσεις, είτε πολυεθνικέ είτε όχι, πρέπει να αναλάβουν σήμερα το μερίδιο της ευθύνης που τους αναλογεί. Μετά από το ατύχημα τη 24 η Απριλίου, βεβαίω κάποιε επιχειρήσει υπέγραψαν συμφωνία για την ασφάλεια. Δεν αρκεί όμως, διότι η πρωτοβουλία αυτή ξεκίνησε πέρσι, χρειάστηκαν όμως άλλοι χίλιοι νεκροί πριν πάρει σάρκα και ωστά. Δεν αρκεί, διότι μόνο άλλωστε ένα τρίτο των επιχειρήσεων υπέγραψε την συμφωνία. Και δεν αρκεί γιατί δεν υπάρχουν και έλεγχοι επιτόπου. Ποια είναι η λύση λοιπόν. Σε ό,τι με αφορά θεωρώ ότι οι επιχειρήσει οι οποίε αναλαμβάνουν την εταιρική του κοινωνική ευθύνη πρέπει να υποχρεωθούν νομικώ να εκπληρώσουν τι υποχρεώσει του. Είναι απαράδεκτο να διεφημίζουν οι επιχειρήσει στην εταιρική κοινωνική ευθύνη και τι καλέ του ενέργειε και από την άλλη μεριά να επιβάλλουν στου υπεργολάβου του συνθήκε οι οποίε δεν του επιτρέπουν ακριβώ να συμμορφωθούν με την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Πρέπει όλα αυτά λοιπόν να γίνουν υποχρεωτικά. Πρέπει να κάνουμε κάτι περισσότερο έτσι ώστε τα λόγια και οι διακηρύξει των επιχειρήσεων να γίνουν πράξει. Κύριε Πίτροπε, είπατε ότι ενδέχεται να αναστείλουμε την ισχύ των προτιμήσεων υπέρ του Μαγκλαντέ στο πλαίσιο του όλα εκτό από όπλα. Δεν νομίζω όμω ότι είναι η κατάλληλη λύση. Πρώτον διότι οι προτιμήσει αυτέ δεν είναι σημαντικέ συγκρινόμενε με το συνολικό όγκο των εξαγών του, του Μπαγκλαντές. Δεν πρόκειται να πιέσουμε έτσι τι αρχέ τη χώρα. Επιπλέον, από την πλευρά μα, χορηγήσαμε κατά εξαίρεση προτιμήσεις για τον τομέα τη φαντουργία ε, στο Πακιστάν και το ίδιο στην ε, Βερμανία. Πιστεύετε, κύριε Επίτροπε, ότι έχει νόημα να στιγματίσουμε το Μπαγκλαντές σε μια στιγμή όπου πλήρεται ταυτόχρονα από φυσικές καταστροφές, πολιτική αστάθεια και ανθρωπινά δράματα. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία συνάδελφος, κύριος Ρέγνα. Ή κυρία Ρέγνα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η κατάρρευση του εργοστασίου στην ΤΑΚΑ είναι μία από πολλές τρομερές τραγωδίες που έχουν προέλθει από τη συστηματική παραβίαση προδιαγραφών ασφαλείας και εργασιακών δικαιωμάτων σε χώρες όπως το Μπαγκλαντές. Πριν από λίγους μήνες είχαμε αντιμετωπίσει μια παρόμοια τραγωδία την πυρκαγιά στο Μπαγκλαντές. Η ευρωπαϊκή αγορά είναι τώρα η κυριότερη αγορά για τα προϊόντα του Μπαγκλαντές που έρχονται ε, σε πολύ φθηνές τιμές χάρη στην δημιουργία επιχειρήσεων πολύ χαμηλής ε, πολύ χαμηλού κόστους που χρησιμοποιούν εργαζόμενους σε απάνθρωπες συνθήκες. Χρειαζόμαστε μια αλυσίδα υπευθυνότητα στην οποία να δεσμεύονται οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Θα πρέπει να έχουμε μια παρακολούθηση και μια έκθεση και ανεξάρτητους ελέγχους σε όλες αυτές τις επιχειρήσεις και την υποχρέωση επανόρθωσης από την πλευρά αυτών των επιχειρήσεων και πάνω απ' όλα χρειαζόμαστε ελεύθερα συνδικάτα τα οποία μπορούν πράγματι να ασκούν τα δικαιώματά τους και όχι να περιορίζονται και να καταστέλλονται. Και θέλω να επαναλάβω αυτή την αίτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να είναι και ένα σημείο επαφής στον Μπαγκλαντές για παράπονα κατά των ευρωπαϊκών επιχείρησεων. Νομίζω λοιπόν ότι είναι μια σαφής η υποστήριξή μας κύριε Επίτροπε προς εσάς, αλλά αναμένουμε να έχετε την απαραίτητη αντιμετώπιση ένα των μεγάλων επιχειρήσεων που έχουν μεγάλη ευθύνη για όλα αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Αρέγνερ. Ο κύριος Φεραίρο έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία, κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η τραγωδία του Μπαγκλατές μας υπενθυμίζει ένα γνωστό πρόβλημα την άκρα εκμετάλλευση και την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις πολυεθνικές που τροφοδοτούν τις ευρωπαϊκές ε, αγορές. Ακόμα χίλιες και πάνω ζωές χάθηκαν στο βωμό του καπιταλισμού. Είναι η χώρα που παράγει πάνω από 90% των κλωστοϊφαντουργικών στον κόσμο και τροφοδοτεί τη ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, τον Καναδά και τις ΗΠΑ σε συνθήκες απάνθρωπες, άθλιες από άποψη υγείας με εργαζόμενους οι οποίοι δεν έχουν καν εργασιακό δικαίωμα και παίρνουν μόνο 30 ευρώ το μήνα. Πάνω από 5.000 βιομηχανίες και εργοστάσια στον χώρο της πρωτεύουσας του Μπαγκλαντές. Πρέπει επιτέλους η Ευρωπαϊκή Ένωση να δράσει εναντίον των επιχειρήσεων που εκμεταλλεύονται αυτή την κατάσταση και αυξάνουν τα κέρδη τους. Να υπάρξουν μηχανισμοί για να αντιμετωπιστούν οι, οι εισαγωγές προϊόντων από αυτές τις περιοχές. Σας ευχαριστούμε κύριε Φεραίρα, ο κύριο σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η καταστροφική κατάρρευση του εργοστασίου στο, στην Τάκα με πάνω από 1.100 ε, νεκρούς και πάνω από 5.000 τραυματισμένους, αυτό κάνει απαραίτητη τη σημερινή συζήτηση. Πολλοί συνάδελφοι τόνισαν ότι υπήρξε μια συμφωνία της προηγούμενης εβδομάδας από 50 διεθνείς επιχειρήσεις κλωστοεφαντουργικών μαζί με ΜΚΟ και εργασιακά συνδικάτα. Πρόκειται όμως και για τις επιχειρήσεις προμήθειας που είναι πάνω από χίλιες για όλες αυτές τις επιχειρήσεις. Θα πρέπει να γίνει γνωστό από πού προέρχονται οι προμήθειές τους θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι και για τους εργαζόμενους στο Μπαγκλαντές θα υπάρχει η απαραίτητη προστασία των εργασιακών συνδικών και των συνδικών ασφάλειας. Πρέπει οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να αναλάβουν επιτέλους την ευθύνη για να τηρούνται οι ελάχιστες προδιαγραφές για τον εξαρισμό, για την πυροπροστασία στις ε, χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας και φυσικά για την σταθερότητα και την ασφάλεια των κτίριων και η Τζιν Λάμπερτ, η οποία είναι η επικεφαλής της ε, αντιπροσωπείας για την Νότια και Νοτιοανατολική Ασία, θα πρέπει να παίξει και αυτή το ρόλο της για να εξασφαλίσει ότι γίνονται τακτικοί έλεγχοι και τηρούνται οι προδιαγραφές. Και φυσικά να σταματήσει αυτή η διαφθορά που σοβεί εκεί. Θα πρέπει οι συμβάσεις του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας να τηρούνται μέχρι κεραίας και να ασκηθεί η κατάλληλη πίεση προς τον τομέα αυτό. Φυσικά Πρέπει να έχουμε προδιαγραφές ασφαλείας και για το περιβάλλον και για τα εργασιακά δικαιώματα. Και όλα αυτά έχουν και ένα τίμημα. Το τίμημα αυτό πρέπει να είμαστε έτοιμοι να καταβάλουμε όταν αγοράζουμε τα προϊόντα αυτό. Αυτό είναι απαραίτητο σε επίπεδο δικαιοσύνης, σε επίπεδο ανθρωπιάς και είναι απαραίτητο να καταδείξουμε τον τρόπο αυτό την ορατή μας αλληλεγγύη. Ευχαριστώ πολύ, ο πρόεδρος, ο κ. Μάρτιν Ντέιβιτ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ευχαριστήσει τον Επίτροπο Ντεκούχτ για την πολύ ξεκάθαρη απάντηση και την ανταπόκρισή της στι τραγωδίε. Υποστηρίζω πλήρω το αίτημα αυτό για τον τελογικό κώδικα και όπω αναφέρθηκε οι εταιρείε που αρνούνται να συμμορφωθούν με αυτόν θα πρέπει να κατονομάζονται. Το μήνυμα που θα πρέπει να πορεύσει από τι τραγωδίε είναι ότι οι πολυεθνικέ αλυσίδε δεν μπορούν να διαφύγουν από τι ευθύνε του μετεγκαθιστώντα τι επιχειρήσει του σε χώρε ή να ισχυρίζονται ότι δεν φέρουν καμία ευθύνη όσον αφορά την όλη αλυσίδα παραγωγή. Ακόμα και αν μπορούν να υπερκεράσουν τον νόμο, δεν μπορούν να ξεπεράσουν την κρίση του κοινού και τι πιέσει που απορρέει από το, οι πιέσει από το κοινό θα τι κάνει αλλάξουν. Και θα πρέπει να υπάρχουν προδιαγραφέ εργασία και να συμπεριλαμβάνονται αυτέ στι συνθήκε, στι συμφωνίε. Θα πρέπει οι αναπτυσσόμενε χώρε να επικυρώσουν και να εφαρμόσουν όλε τι προδιαγραφέ για το χώρο εργασία και καλωσορίζω την απόφαση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξεκινήσει έρευνε όσον αφορά το πόσο συμμορφώνεται με τι με τις προδιαγραφέ τη γενικευμένη προτιμής των Μπαγκλαντέ. Δεν πρόκειται περί τιμωρία που θα επιβληθεί στο Μπαγκλαντέ. Θέλουμε να ενθαρρύνουμε τον Μπαγκλαντέ να βελτιώσει συνθήκε εργασία στου εργαζομένου και οι προδιαγραφέ υγιεινή και ασφάλεια να είναι σε υψηλό επίπεδο και προστατεύονται τα δικαιώματα των εργαζομένων. Δεν θέλουμε να τιμωρήσουμε τον Μπαγκλαντέ. Θέλουμε να ενθαρρύνουμε τον Μπαγκλαντέ να ακολουθήσει καλύτερο μονοπάτι. Ευχαριστώ. Thank you. Thank you very much. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Τούσας έχει το λόγο τώρα. Η τραγωδία κατάρρευσης του οκταόροφου κτηρίου που στέγαζε βιοτεχνίες ενδυμάτων στα κάτεργα της Ράνα Πλάζα στο Μπαγκλαντές και οδήγησε στο θάνατο πάνω από χίλιους εργάτες αποτελεί κρίκο στην αλυσίδα των αμέτρητων εγκλημάτων του καπιταλισμού σε βάρος της εργατικής τάξης. Όπως αυτά που συμβαίνουν καθημερινά κατά χιλιάδες στις καπιταλιστικές χώρες, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη ΣΥΠΑ, την Ιαπωνία και άλλες και βαφτίζονται προκλητικά εργατικά ατυχήματα η εργοδοτική τρομοκρατία η εντατικοποίηση της δουλειάς οι ελαστικές μορφές απασχόλησης με 12 έως 16 ώρες δουλειά την ημέρα κατά την περίοδο αιχμής της παραγωγής σε επικίνδυνες υποδομές στους χώρους δουλειάς χωρίς κανένα έλεγχο προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η κερδοφορία των μονοπωλίων αποτελούν τις βασικές αιτίες των τραγικών εργατικών ατυχημάτων. σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του διεθνούς οργανισμού εργασίας ένας εργαζόμενος ανά τρία λεπτά χάνει τη ζωή του από εργατικό ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια. οι προτάσεις του κοινού ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων του ευρωκοινοβουλίου που καλεί τους καπιταλιστές να εφαρμόσουν την εταιρική κοινωνική ευθύνη δηλαδή να ελέγχουν οι ίδιοι τον εαυτό τους αποσκοπούν να διαιωνίσουν την καπιταλιστική βαρβαρότητα της εκμετάλλευσης εργατικής τάξης αποτελούν πρόκληση για τους συγγενείς των θυμάτων και την εργατική τάξη συνολικότερα. μόνο οι οργανωμένοι πάλι μέσα στους τόπους δουλειάς μπορεί να επιβάλλει να ληφθούν μέτρα για την προστασία των εργαζομένων μπορεί να ανατρέψει αυτό το σάπιο καπιταλιστικό σύστημα την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο την κατάργηση της εργατικής λαϊκής εξουσίας. Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ συνάδελφοι. Έχετε ξεπεράσει κατά 50% το χρόνο σας. Πρέπει όμως να εξασφαλίσω την ισότητα μεταξύ των ομιλητών. Ο κύριος Κέλλη. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Όσον αφορά λοιπόν το θέμα αυτό, συνάδελφοι, θα πρέπει να εκφράσω και εγώ τα συλληπιτήριά μου προς τους, ε, στο λαό της Βρετανίας για αυτό που συνέβη στους δρόμους της. Αυτό που συνέβη στο Μπαγκλαντές δεν χρειαζόταν να συμβεί. Οι επιθεωρητές είπαν την προηγούμενη ημέρα ότι το εργοστάσιο δεν ήταν ασφάλες ε, και παρόλα αυτά οι ιδιοκτήτες του εργοσταρίου πίεσαν τους εργαζομένους να μπουν και ξέρουμε ποιο είναι το αποτέλεσμα. Πάνω από χίλιοι σκοτώθηκαν. Δεν χρειάζεται να συμβαίνει αυτό. Δεν θα έπρεπε να το ανεχθούμε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αγανάκτηση υπάρχει για αυτό που συνέβησαν στον Μπαγκλαντές και σωστά ο Πάπας είπε ότι αυτό που το συνεγγνώρισε περισσότερο ήταν ότι πληρωνόταν 30 ευρώ το μήνα αυτοί οι εργάτες και θεώρησε ότι αυτό είναι δουλεία και σωστά το είπε. Και το κέρδος θεώρησε ότι μπαίνει πάνω από τον άνθρωπο και εκεί έχει δίκιο. Ε, έχουμε λοιπόν υποχρέωση να προσπαθήσουμε να το αλλάξουμε αυτό και νομίζω ότι έχει δίκιο Ευρω... ο επίτροπο, και όπω είπε η Ρίζα Πεθκόστιγκερ λέω και εγώ ότι πρέπει να είμαστε πρεσβευτέ για τι προδιαγραφέ τις ευρωπαϊκές θα πρέπει να συνεργαστούμε με τι αρχέ του Μπαγκλάντε, να εξασφαλίσουμε τα ύψιστα πρότυπα που θα πρέπει να ισχύουν και τα κτίρια θα πρέπει να καταδικάζονται ως αχρησιμοποίητα και να μην μπορούν να υποχρεώσουν οι ιδιοκτήτε των κτιρίων να, να υποχρεώσουν τον κόσμο να μπει να δουλέψει εκεί. Θα πρέπει να του βοηθήσουμε να εξετάσουν και άλλα ατυχήματα τα οποία ίσως θα μπορούσαν να συμβούν για να αποφευθεί κάτι παρόμοιο. Και τέλος, οι μεγάλες πολυεθνικές του Λιανικού πρέπει να υποχρεωθούν, υπογράψουν δεντολογικό κώδικα και αν δεν το κάνουν να ζητήσουμε από το κοινό να μην υποστηρίζει τα αγαθά τους. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Μπάτια Ικουτσέτ. Έχει το λόγο κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Και εγώ θέλω να προσθέσω τα δικά μου συλληπιτήρια προς τις οικογένειες των θυμάτων αυτού του τρομερού ατυχήματος που έλαβε χώρα στο εργοστάσιο του Μπαγκλαντές. Εκφράζω τη λύπη μου για τις επισφαλείς συνθήκες εργασίας στις οποίες εργάζονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι και την απάθεια και την έλλειψη εφαρμογής των κανόνων που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια στον χώρο εργασίας που είναι και η πηγή αυτού του ατυχήματος και επίσης θέλω να καταδικάσω και την ατιμορρησία των ιδιοκτητών αυτών των εργαστοσίων, όπου έχουν γίνει αυτά τα τρομερά ατυχήματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επειδή είναι ο κύριος ε, χώρος διάθεσης αυτών των προϊόντων από τον Μπαγκλαντές θα πρέπει να δράσει για να εμποδίσει την επανάληψη αυτών των φαινομένων. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλους τους μηχανισμούς που είναι στη διάθεσή μας και να εξαρτήσουμε και την ελεύθερη πρόσβαση των προϊόντων αυτών στην ευρωπαϊκή αγορά από την ε, πλήρη τήρηση των διεθνών συμβάσεων για τα εργασιακά δικαιώματα και την ασφάλεια στον χώρο εργασία. Χαιρετίζω το γεγονό ότι κάποιε από τι εταιρείε αυτέ έχουν ήδη ε, δεχτεί τη συμφωνία για την ασφάλεια και επίση χαιρετίζω και τι προσπάθειε του Μπαγκλαντέ να μεταρρυθμίσει τι ε, συνθήκε εργασία τη επιχειρήση. Δεν πρέπει όμω να σταματήσουμε εδώ, θα πρέπει να συνεχίσουμε να παίζουμε ένα προορατικό ρόλο στο να εξασφαλιστούν οι αρχές της εταιρική υπευθυνότητας και θα πρέπει να προωθήσουμε μια καλύτερα πληροφορημένη μορφή κατανάλωσης, μια καλύτερη ετικετοθεσία που καταδεικνύει ποιες επιχειρήσεις πράγματι τηρούν όλα αυτά τα κριτήρια και γι' αυτό επικροτώ και τις, προσπά... προτάσεις που μας έχει κάνει η Κομισιόν και ελπίζω ότι θα μπορέσουν πράγματι να εφαρμοστούν. Ευχαριστώ. Ο κ. Κομφεράτη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αυτό που συνέβη στη Ράνα Πλάτζα είναι ένα δράμα που θα μπορούσε να το προβλέψει κανείς πάρα πολύ εύκολα και που συνέβη εν τη αδιαφορία του μεγαλύτερου ποσοστού των πλουσίων χωρών που γνωρίζουν ότι υπάρχουν αυτές οι συνθήκες που παράγουν με στόχο τη συγκράτηση του κόστους χωρίς να βλέπουν ποιες συνθήκες ε, εργάζονται τα άτομα που ασχολούνται με, αυτό, με αυτή την παραγωγή. Τα δικαιώματα τη εργασία είναι θεμελιώδη σε οποιοδήποτε μέρο του κόσμου. Αλλά έχουμε μια σοβαρή ευθύνη και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να δράσουμε τάχιστα. Δεν μπορούμε να ανεχθούμε ακόμα συνθήκε αυτού του είδου. Έχουμε τα κατάλληλα εργαλεία για να κινηθούμε αρκεί να συμπεριληφθούν σε συμφωνίε, συμφωνίες, να μπει μια ρήτρα που δεσμεύει τι χώρε και τι επιχειρήσει που λειτουργούν στι χώρε αυτές να σέβονται τι συνθήκε τη στοιχειώδης που αφορούν του εργαζομένου. Αρκεί λοιπόν να προάγουμε κυρώσεις ε, απέναντι στις ευρωπαϊκές εταιρείε που δεν σέβονται τις οδηγίες ε, του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας. Εμείς λοιπόν ε, δεν είμαστε διαφορετικοί από τον υπόλοιπο κόσμο. Είμαστε οι κύριοι χρήστες και γι' αυτό το λόγο έχουμε μια ηθική υποχρέωση να προστατεύουμε τους υπόλοιπους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περνάμε λοιπόν τώρα στη διαδικασία Catch the Eye και έχουν ζητήσει εννέα αγορητές το λόγο. Επειδή λοιπόν έχουμε αρκετό χρόνο στη διάθεσή μας, θα δώσω το λόγο και στους εννέα. Και ξεκινάμε την κυρία Πρενταγκάστ. Σας ευχαριστώ πολύ. Επειδή το Μπαγκλαντές είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος το Ηνωμένο Βασίλειο δεν μπορεί να μένει αδιάφορο. Το Διεθνές Γραφείο Εργασίας ε, έχει αρχίσει τις ε, ε, προβλέψεις και τις ενέργειες για το τι συμβαίνει στον κόσμο της εργασίας σε αυτή τη χώρα. Το κτίριο αυτό είχε εντοπιστεί σε προγενέστερη φάση πριν καταρρεύσει το Μπαγκλαντές λοιπόν ε, δεν έχει ειδική μεταχείριση υπάρχει βέβαια κάποιο σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει οικονομική ανάπτυξη αλλά πρέπει να προστατεύονται και οι ζωές των εργαζομένων και να διασφαλίζονται αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας ως ε, μεμονωμένοι καταναλωτές ε, ε, δεν πρέπει να δεχόμαστε αυτές τις συνθήκες της κατασκευής και παραγωγής ενδυμασίας και ρούχων. Πρέπει λοιπόν να γίνονται σεβαστές οι διατάξεις του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας που αφορούν σε αυτές τις εταιρείες. Πρέπει να εφαρμόσετε μια κοινωνική πολιτική. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η κυρία Αντρές Παρία έχει το λόγο. Έχουμε πάνω από 1100 θανάτου σε αυτό το εργοστάσιο στον Πελαντέ. Αυτό είναι απαράδεκτο, είναι μια ντροπή. Οι συνθήκε εργασία, η κατάσταση των εργαστών κλπ. Και εμεί είμαστε οι πρωταθλητέ όσον αφορά την εισαγωγή των κλωστοματουργικών. Αυτό ε, επιπλέον, λόγω τη κερδοσκοπία που γίνεται όσον αφορά του χαμηλού μισθού, βλάπτει και τι δικέ μα ε, εξαγωγέ. Οπότε αυτό το οποίο πρέπει να γίνει είναι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να, ε, να, να κατοχυρώσει το δικαίωμα αυτό ε, θα πρέπει να τι θα σέψει τις ε, πολυεθνικές έχουμε 24 τέτοιες που δρουν εκεί και έχουμε ένα σωρό άλλες οι οποίες αγοράζουν προς από τον Παγκλαντές και επομένως αυτοί οι οποίοι λένε ότι αυτά είναι μικρές ποσότητες θα πρέπει να πειθαρχίζουν εκείνους ορμόνες οι οποίοι δεν συμμορφώνονται με τις ε, διατάξεις του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας. Έχουμε πάρα πολλά τέτοια την οποία έχουν γίνει. Η κυρία Μιράντα, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η τραγωδία αυτή δείχνει την ε, ολιγορία. Είναι πάρα πολύ ε, ε, χτυπητό παράδειγμα προς αποφυγή γιατί μιλάμε τώρα για εκμετάλλευση του φτωχού και έχουμε πάρα πολλούς οι οποίοι σκοτώθηκαν εκεί είναι το Μαγκλαντές στη δεύτερη θέση του, των εξαγωγέων ε, παγκοσμίω για τα κλωστοβαντουργικά και τα, και τα ενδύματα. Επομένως θα πρέπει να υλοποιηθούν όσα προβλέπονται για την ευθύνη στο διεθνές εμπόριο και θα πρέπει να κάνουμε κάτι για αυτές τις γυναίκες που δουλεύουν σε αυτόν τον κλάδο και έχουν πάρα πολύ χαμηλούς μισθούς, έχουν συνθήκες εργασίας ε, πάρα πολύ κακές, ε, βάλωθες δουλεύουν ε, υποπίεση, επομένως είμαστε όλοι υπεύθυνοι και εμείς που καταναλώνουμε τα προϊόντα αυτά. Και η προηγούμενη επιτροπή δεν έκανε τίποτα όταν είχαν πρώτα αναφύγει αυτά τα ζητήματα. Χρειάζεται επομένω να κάνουμε κάτι όσον αφορά μια, μια δεσμευτική κοινωνική ευθύνη των εταιριών. Κυρία Γιακονσάρη, παρακαλώ. Ε, ε Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω. Toinen tärkeä asia on se, että me Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη σαφέστατη θέση που έλαβε. Αυτό που έχει σημασία είναι το εξή, ότι ε, θα πρέπει να ε, ταχθούμε υπέρ αυτών των νομοθετικών μέτρων που προστατεύουν τους εργαζόμενους. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η ε, παρουσία προς τα έξω και η διαμόρφωση κοινή γνώμης είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Μόνο με τον τρόπο αυτό μπορούμε να κάνουμε σωστό έλεγχο. Βεβαίως αυτό είναι και ένα θέμα του ρόλου των γυναικών. Αν δούμε την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή, ε, αν, στην περίπτωση κατά την οποία προκύπτει ένα μικρό ατύχημα, στις ε, ειδήσει ε, εμφανίζεται το ατύχημα αυτό. αν στο ατύχημα αυτό επλήττονται μόνο γυναίκες, τότε τα μέσα ενημέρωσης δεν θα το προέβαλαν. Γνωρίζουμε βέβαια ότι και οι καταναλωτές φέρουν μια κάποια ευθύνη. Οφείλουμε να ξέρουμε τι ακριβώς παράγουν αυτά τα εργοστάσια. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε και κύριοι. Καταρχήν θα ήθελα να εκφράσω την απογοήτευσή μου για το ότι δεν είναι πλέον εδώ ο Επίτροπος κύριος Ντεκούχτ, διότι σε τελική ανάλυση ε, πήρε την δική μας την σύμφωνη γνώμη παλαιότερα, όταν είχαμε το παλαιότερο ατύχημα, ε, όπου είχαμε πει ότι οι γενικές προτιμήσεις θα πρέπει να εφαρμόζονται για να προστατεύουν καλύτερα τα εργοστάσια. Ε, θα ήθελα, θα προτιμούσα να ακούσω τη συζήτηση μέχρι τέλους και μετά να εκφράσω τα δικά μας τα αιτήματα. Ένα αίτημα δικό μας είναι η γερμανική πρεσβεία αλλά και άλλοι φορείς να δέχονται τις διαμαρτυρίες ε, και να τις μεταφέρουν. Αλλά σε επανέλθουμε στο θέμα μας. Πρέπει κάθε φορά να πεθαίνουν, να χάνουν τη ζωή τους εκατοντάδες άνθρωποι πριν σοκαριστούμε για να θεσπίσουμε τα απαραίτητα μέτρα. Βεβαίως και όλους, όλους μας αρέσουν τα ωραία ρούχα, τα μοντέρνα ρούχα, όμως πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Ε, θα πρέπει να μην δεχόμαστε να μην αγοράζουμε ε, ρούχα από εταιρείε όπω από την ΚΑΠ και από άλλε που κατασκευάζουν τα ρούχα σε αυτές τις ε, χώρε να του πούμε κοιτάξτε να προστατεύετε καλύτερα του εργαζόμενου, να εφαρμόζετε ε, μέτρα προστασία, πυροπροστασίας και να επιτρέπετε και το συνδικαλισμό. Να πω ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε και τι μη κυβερνητικέ οργανώσεις οι οποίε εδώ και δεκαετίε αγωνίζονται για να βελτιωθούν οι συνθήκε εργασία για να γίνεται σεβαστή η αξιοπρέπεια των εργαζομένων στα εργοστάσια αυτά. Ευχαριστούμε. Κύριος Μέρφυ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Πράγματι η εργασία είναι ευθυνή αλλά και η ζωή είναι ευθυνή για εκατομμύρια εργαζομένων στην βιομηχανία της ένδυσης στο Μπαγκλαντές. Τέσσερα εκατομμύρια από τα οποία οι περισσότεροι γυναίκες. Μετά από την τελευταία καταστροφή άνω των χιλίων νεκρών για την εξυπηρέτηση του, ε, ε, αυτού του καπιταλιστικού απαιτητικού συστήματος. Gap, Metro, Walmart έχουν κερδίσει πάρα πολλά από την ευθυνή αυτή μορφή εργασίας ε, και κερδίζουν 3 με 5% από την τελική τιμή. Αλλά για να εκμεταλλευτούν ακόμα περισσότερο τους εργαζομένους ε, ε, καταστέλουν τα συνδικαλιστικά δικαιώματα. Λόγω της ε, κατακραυγής των τελευταίων ημερών κάποια βήματα έγιναν αλλά παρόλα αυτά όλα αυτά εκθέτουν θα έλεγα ε, την ε, υποκριτική πλευρά των λεγόμενων προγραμμάτων εταιρικής υπευθυνότητας ή κοινωνικής υπευθυνότητας των εταιριών. Αν πρέπει να σταματήσει η εκμετάλλευση θα πρέπει να φύγουν τα εργοστάσια από αυτούς που παράγουν αποκλειστικά για το κέρδος και να περάσουν στον έλεγχο των ιδίων των εργαζομένων. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Μετά την τελευταία καταστροφή ε, στο Μπαγκλαντές ε, πρέπει να εφαρμοστεί μια σειρά μεταρρυθμίσεων από διατάξεις ασφαλείας μέχρι τον κατώτατο των μισθών και τον συνδικαλισμό. Όλα αυτά πρέπει να βελτιωθούν. Βεβαίως ε, κατά πόσον θα ακολουθήσουν συγκεκριμένα δεδομένα όσον αφορά αυτά θα δούμε. Υπάρχουν κακές συνθήκες εργασίας οι οποίες βέβαια δεν περιορίζονται μόνο στο Μπαγκλαντές. Αυτό το γνωρίζουμε και δεν αφορούν μόνο τον τομέα μην ξεχνάτε τι συνέβεται πρόσφατα που κατέρευσε η οροφή ενό εργοστασίου στην Καμπότζη. 37 ε, διεθνεί οργανώσει ε, έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Πυροπροστασία στο Μπαγκλαντέ και αυτό θα μπορούσε να αποτελεί μια σημαντική αλλαγή. Αν αυτό βέβαια μπορεί να εφαρμοστεί ε, στην πράξη θα ήταν ακόμα καλύτερο και να αφορά όχι μόνο τι ευρωπαϊκέ εταιρείε, αλλά και τι αμερικανικέ. Προ αυτή την κατεύθυνση πρέπει να εργαστούν και οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί δεν είναι δυνατόν οι πολυεθνικές εταιρείες να ασκούν πίεση στις χώρες ευθυνής παραγωγής απλά και μόνο για να μεγιστοποιούν το κέρδος τους. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Ιρεγκόιαν Πέρες έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Από ό,τι αφορά τιμή στα θύματα του Μπαγκλαντές, πρόκειται για αυτή το, το, το, την κοντόφθαλμη άποψη που έχουμε εδώ από την Ευρώπη θα πρέπει να μπορέσουμε κάτι να κάνουμε για να σταματήσει αυτή η εκμετάλλευση, αυτή η κατάσταση της ε, δουλείας, όλα αυτά που έχουν καταδικαστεί από τον ΟΗΕ, αυτοί οι άνθρωποι που παίρνουν λιγότερο από 30 ευρώ το, το, το μήνα, όλα αυτά είναι απαραίτητα σε καταστάσεις αναξιοπρεπείς, επομένως πρόκειται για παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων ε, αυτών των ανθρώπων και έστω για να από τρίτε χώρε θα πρέπει να εφαρμόζονται και για αυτού αυτό που θέλουμε και για τον εαυτό μα. Επομένω, θα πρέπει να προσέχουμε τι διεθνέ μα σχέσει και να ε, προσέξουμε, προστατεύσουμε αυτούς οι οποίοι έχουν τα ρούχα που φοράμε. Θα πρέπει κάτι να κάνουμε για την κοινωνική ευθύνη. Δεν ωφελούν οι καλές πρακτικές. Θα πρέπει να ισχύσουν οι κανόνες του ΩΣΑ, του Γραφείου Εργασία και του ΠΟΕ, να παράσχουμε κάποιες ευθύνε για ασφάλεια, για αξιοπρέπεια και για προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων. Επομένως, τίποτα παραπάνω από το να τηρούνται τα όσα έχουν συμφωνηθεί. Η κυρία Γιατιμάκη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Χίλιοι νεκροί λοιπόν στο Μπαγκλαντές, μια πραγματικά τεράστια τραγωδία. Η βασική ευθύνη για την ε, τραγωδία αυτή φυσικά ανήκει στους ιδιοκτήτες του κτηρίου και στις αρχές, τις ελεγκτικές της συγκεκριμένης χώρας. Έχουμε και εμείς όμως ευθύνη εμείς θα πρέπει να γνωρίζουμε από πού προέρχονται τα εμπορεύματα που εισάγουμε. Θα πρέπει τα εμπορεύματα αυτά να είναι ασφαλή και να μην βλάπτουν τους πολίτες. Και δεν γνωρίζουμε πώς λειτουργούν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και οι υπεργολάβοι τους στις χώρες του τρίτου κόσμου. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δράσει, να μην μας ενδιαφέρει μόνο το θέμα της ασφάλειας των προϊόντων, το οποίο είναι σημαντικό, αλλά να δούμε ακριβώς τις συνθήκες παραγωγής, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για προϊόντα που ανήκουν και παράγοντα από ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ε, κλείνουμε λοιπόν με τον κύριο Περέλο Ροντρίγκε. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αυτό το οποίο συνέβη στον Παγκλαντές δεν είναι ένα ατύχημα. Είναι η συνέπεια όλων αυτών των ετών που επιτρέπεται όλοι αυτοί να κερδίζουν κόντρα σε κάθε αρχή ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κοινωνικής δικαιοσύνης, συνθήκων και, και προστασίας των εργαζομένων. Και επομένως αυτό το οποίο χρειάζεται δεν είναι τα, τα ψηφίσματα, είναι να υπάρξει μια καινούργια ηθική στις επιχειρήσεις. Έχουμε ικανός αρκετούς μηχανισμούς ούτως ώστε να επιβάλλουμε αυτήν την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Κάποια μέτρα που να ξεκαθαρίζουν και να φαίνεται ποιος τα εφαρμόζει, ποιος δεν τα εφαρμόζει, ποιος εφαρμόζει συνθήκες δουλειέ και ποιος όχι. Να είναι αυτό γνωστό και να προβάλλεται αυτός ε, ο οποίος είναι παρόν προ μίμηση και αυτό να προβάλλεται και στους καταναλωτέ. Ε, από σε ψήγμα πάμε, αλλά αυτό δεν ωφελεί. Θα πρέπει τα λόγια να γίνουν έργα, αν θέλουμε μια αξιοπρεπή Ευρώπη με αξιοπρεπείς Ευρωπαίους που αυτό που καταναλώνουν επίσης είναι αξιοπρεπές. Άρα θα πρέπει να κάτσουμε και να εξελογήσουμε τα πράγματα για να αποφύγουμε την ομαλέψη τέτοιων τραγωδιών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ε, θα ήθελα να σας παρακαλέσω στο μέλλον να μιλάτε λίγο πιο αργά, λέει ο Πρόεδρος, γιατί δημιουργείται προβλήματα στη διερμηνία όταν μιλάτε τόσο γρήγορα. Και τέλος ε, θα απαντήσει ο Επίτροπος κύριος Ότιγκερ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί κυρίες και κύριοι βουλευτές, συμφωνούμε ως προς την αξιολόγηση των τραγικών γεγονότων και βεβαίως και είμαστε συγκλονισμένοι. Ο συνάδελφός μου, κύριος Εντεγκούχτ, ε, ο οποίος ε, έκανε την ανάλυση και κατέδειξε ποια μέτρα ε, θα λάβει εκείνο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν δυστυχώς αναγκασμένος να επιστρέψει στις Βρυξέλλες επιγόντως. με παρεκάλεσε να τον αντικαταστήσω. Είναι παρόν οι εκπρόσωποι του πολιτικού του γραφείου και θα του μεταφέρω κι εγώ. αυτά τα οποία λέτε βρίσκουν τη συγκατάθεσή μας. Ο συνάδελφος ε, κύριος Ντεγκούχτ, ε, το ακούσατε, ε, συμφωνεί με αυτά που είπατε κι εσείς. Δεν υπάρχει αντίφαση μεταξύ αυτών που είπε ο κύριος Ντεγκούχτ και μεταξύ των δικών σας παρατηρήσεων. Οι επαφές με την κυβέρνηση του Μπαγκλαντές έχουν αναλυφθεί με τον Πρωθυπουργό, με τους αρμόδιους υπουργούς και η συνεργασία ε, καταρχήν είναι το πιο σημαντικό μέτρο ε, η συνεργασία με την κυβέρνηση. Μετά θα προχωρήσουμε σε συνεργασία με τις ε, βιομηχανίες και τις πολυεθνικές εταιρείες οι οποίες οφείλουν να ενημερώσουν και τις, τους προμηθευτές τους. Πράγματι αυτό που πρέπει να ζητήσουμε είναι να υπάρχουν ελάχιστες προδιαγραφές για την προστασία της εργασίας, για τις συνθήκες της εργασίας, για την πυροπροστασία, για την ασφάλεια των κτηρίων. Ε, πρέπει να τηρούνται οι κοινωνικές ε, προδιαγραφές, ε, προδιαγραφές εργασία που ισχύουν σε ολόκληρο τον κόσμο. Θα συνεχίσουμε τη συνεργασία μας με το Διεθνές Γραφείο Εργασίας και μπορείτε επίσης να θεωρήσετε βέβαιο το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μεριμνά για την τήρηση αυτών των προδιαγραφών ανεξάρτητα με το που παράγονται τα προϊόντα το γεγονός ότι είμαστε συγκλονισμένοι, όπως σας είπα αυτό θα οδηγήσει σε συγκεκριμένες πράξεις. Ο συνάλφος κύριος Ντεγκούχτ έχει ήδη κάνει τα πρώτα βήματα έτσι ώστε έστω και εκ των υστέρων να συμβάλλουμε και εμείς στη βελτίωση των συνθήκων εργασίας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις επικοδομητικές σας προτάσεις που θα μας βοηθήσουν στο έργο μας. Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και Έξι προτάσεις ψηφίσματος κατατέθηκαν. Κατόπιν τούτου ολοκληρώνεται η συζήτηση και η ψηφοφορία θα λάβει χώρα αύριο, αύριο στις 12 ε, μάλλον εκ παραδρομής αύριο είπε ο Πρόεδρος. Θα λάβει χώρα στις 12. Να ρωτήσω τον Επίτροπο Έτιγκερ κάτι. Δεν ξέρω αν άκουσε αυτό που του είπα. Συνάδελφε, έχει ολοκληρωθεί η συζήτηση. Η ψηφοφορία επ' αυτού του θέματος ε, δεν λαμβάνει χώρα τώρα. Έκλεισα τη συζήτηση. Αύριο, λέει πάλι ο πρόεδρος εκ παραδρομής,